μπορούν οι βουλευτές ε, να ζητήσουν ως αύριο 17 Απριλίου να αμφισβητήσουν την ε, έναρξη των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να εγκριθεί από την Ολομέλεια μια τέτοια αντίρρηση. βάλλος οι αρμόδιες επιτροπές θα προχωρήσουν στις διαπραγματεύσεις τους βάσει του άρθρο